ich erkläre die 12. September. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση που διακόπηκε στις 12 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σα παρακαλέσω να τηρήσουμε ενό λεπτού σιγή.